αύριο 5η 19 Φεβρουαρίου στις 9 και επιτέλους μπορούμε να σβήσουμε τα φώτα και να λύσουμε τη συνεδρίαση. Καληνύχτα σας.